και ούτε Σαμποτέρο από τις 26 Απριλίου εξελ... εξελέγησαν ε, στο Κοινοβούλιο της Φιλανδίας τους συγχαίρουμε βεβαίως σύμφωνα με το άρθρο 7.2 του κανονισμού αυτό σημαίνει πως είναι πλέον ασυμβίβαστη η ιδιότητα του Εθνικού Βουλευτή με του Ευρωβουλευτή και άρα